Okay, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Συγκάλεσα τη συνεδρίαση αυτή για τους εξής τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή η Επιτροπή Απασχόλησης δεν είχε συγκροτήσει σε σώμα, η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών δεν μπορούσε ούτε εκείνη να συγκροτηθεί σε σώμα. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο ε, το χρονοδιάγραμμα για την ακρόαση των δύο νέων επιτρόπων. Και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών επρόκειτο να συγκρατηθεί σε σώμα την επόμενη Τρίτη. Δεύτερον, αν δεν σε σώμα η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη μας τακτική συνεδρίαση η οποία έχει προγραμματιστεί για την άλλη Τετάρτη. Ας πούμε, ε, στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση του προγράμματος της Φιλανδικής Προεδρίας. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε σημαντικά θέματα ε, πήγοντα να διεκπαιρεώσουμε και αν θέλουμε να έχουμε λόγο ως Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ας πούμε, στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τα δημοσιονομικά, ε, θα είχαμε πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν θέματα προγραμματισμού, χρονοδιαγράμματος για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τα δημοσιονομικά. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θεώρησα επίγον και απαραίτητο να βρούμε μια λύση για να συγκροτηθούμε σε σώμα. Συγγνώμη που δεν σας ρώτησα όλους πριν συγκαλέσω αυτή τη συνεδρίαση, αλλά χτες το βράδυ αργά έμαθα ότι είχαμε βρει αίθουσα και διερμηνία και άδραξα την ευκαιρία. Και χαίρομαι που ήρθατε. Ε, το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Κάζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εξελέγει κοσμήτορ πριν από λίγες μέρες, δύο εβδομάδες. Άρα θα είμαι για τελευταία φορά σήμερα εδώ ε, ως συντονιστής ε, του ΕΛΚ. Φυσικά θα παραμείνω, αλλά όχι ως συντονιστής. Μέλος θα παραμείνω, ε, είμαι κοσμήτρο πια. Και ελπίζω ο κύριος Ντένις Χάτχη να με αντικαταστήσει ως συντονιστή. Εχθές ήταν μοναδική ευκαιρία Ήταν βέβαια ένα σφάλμα αυτό ε, ελπίζω να μην επαναληφθεί, να μην συμβαίνουν πολύ συχνά. Ήταν πραγματικό σφάλμα, αλλά ελπίζω στο μέλλον να υπάρχει διαβούλευση με όλους τους ε, συντονιστές. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει επιγόντως να συγκροτηθούμε σε σώμα και όπως είπε η Άγνες έχουμε σημαντικά θέματα να διεκπαιρεώσουμε. εύχομαι σε όλους όσοι θα εκλεγούν σήμερα καλή τύχη και σε όλους τους συντονιστές ήταν τα καλύτερα πέντε χρόνια, στα 15 χρόνια που είναι με μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ. Εργαστήκαμε πραγματικά ως ομάδα και ελπίζω και οι νέοι συντονιστές να συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία. Δεν θα συμφωνούν πάντα για όλα, προφανώς, αλλά την τελευταία πενταετία λειτουργήσαμε ως ομάδα και ήταν ε, καθοριστικά αυτά τα πέντε χρόνια, πολλά πετύχαμε. Σας εύχομαι άλλη τύχη, καλή επιτυχία και πολύ σκληρή δουλειά για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Επιτροπή μας, που είναι, όπως λέω και εγώ πάντα, από τις σημαντικότερες ε, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και τη χθεσινή ιδιαίτερα, γιατί επικοινώνησα με τους περισσότερους από εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα των συντηρητικών και των μεταρρυθμιστών που έδειξαν κατανόηση για την πολύ δύσκολη κατάσταση και ελπίζω τώρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία γιατί ξέρω ότι αδειμονείτε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you, Mr. Uh, σας ευχαριστώ κύριε Κάσα και σας ευχαριστώ για την uh, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και θα ήθελα να πω και στους υπόλοιπους συναδέρφους ότι πριν από λίγο ζήτησα συγγνώμη για τα τόσο εσπευσμένα συνεκάλεσε αυτή τη συνεδρίαση. Το δηλώνω και πάλι, ζητώ συγγνώμη, θα έπρεπε να είχα ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι και δεν εκτιμώ τη συνεργασία μας και δεν προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία και με τον κύριο Ράτκε και με τους υπόλοιπους συντονιστές. Και αν καταφέρουμε τελικά να συγκροτήσουμε σε σώμα την Επιτροπή Απασχόλησης, μπορούμε να μείνουμε ε, ικανοποιημένοι και να ξεκινήσουμε από τώρα το έργο μας. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε όλες διερμηνίες, όλες τις γλώσσες, που είναι αξιοσημείωτο πράγμα παρόλο που τελευταία στιγμή οργανώσαμε ε, την συνεδρίαση. Δυστυχώ δεν έχουμε Μαλτέζικα, λυπάμαι κύριε Κάζα, και σλοβενικά. Ε, Όλε οι υπόλοιπε γλώσσε όμω ε, υπάρχουν για ερμηνεία. Ή μάλλον όχι, συγγνώμη. Μαλτέζικα δεν έχουμε. Σλοβενικά, δανέζικα, τσεχικά, μόνο παθητικά σλοβενικά, δανέζικα, τσεχικά, μόνο παθητικά. Μπορείτε να μιλάτε δηλαδή, όχι να ακούτε. Επίσης, ε, για τους αντικαταστάτες, εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Κίτενταλ αντικαθιστά τον κύριο Φούρλα, τον κύριο Φούρλα, εκ μέρους των σοσιαλιστών, τον κύριο Φουρλά, συγγνώμη, ε, η κυρία Σαμπίλα, τον κύριο Φλούξαμ, τον κύριο Φούγκελζανκ και από το Ρινιού η Άννα Τζούλια Ντονάτες ε, αντικαθιστά το Τζέιμς Μπρόντι. Από τους Πρασίνους ο Σπάρτακ ε, αντικαθιστά τον κύριο Τατζάνας παρόλο που την είδα στην αίθουσα και από ε, τους, το ID η Σιμώνα Μπαλτάσαρα αντικαθιστά τη Στεφανία Σαμπέλη και από την ΚΟΕ Ο κύριος Πότιγκερ αντικαθιστά μάλλον την κυρία Περέιρα, γιατί πρέπει να μιλήσει στην Ολομέλεια, οπότε θα μπαινοβγαίνει στην συνεδρίαση. Με αυτές τις αντικαταστάσεις λοιπόν που σας ανήγγυλα, μπορώ να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης. Ε, σκοπός της σημερινής μας συνεδρίασης είναι να συγκροτήσουμε σε σώμα το Προεδρείο εκλέγοντας Πρόεδρο και μέχρι τέσσερις αντιπροέδρους. Με τη σειρά που σας ανήγγειλε και στην προηγούμενη συνεδριάση. Πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο και μετά τους τέσσερις αντιπροέδρους. Απαρτία έχουμε και σας ευχαριστώ πραγματικά που ήρθατε. Καταρχήν, ποιοι είναι οι υποψήφοι για τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής ΕΜΠΛ. Η κυρία Ραφάλσκα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εκ μέρους του ECR θα ήθελα να προτείνω ε, για την Προεδρία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων την κυρία Ντουρίση Νικόλσονόβο. Okay, thank you. Thanks for this nomination. Σας ευχαριστώ για την υποψηφιότητα. Οπότε, ερωτώ την υποψήφια δέχεται την, ε, το διορισμό της. Ναι, κυρία Σόνοβα δέχεται την υποψηφιότητα. Κάποιος ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Εκ μέρους ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να ζητήσω διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Μάλιστα, ελπίζω να έχετε όλοι μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας ή τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα. Έχει διαφορά αν ψηφίσουμε κανονικά ή μυστικά. Καλύτερα να κάνουμε τη δοκιμαστική μυστική ψηφοφορία. Και η πράσινη είναι υπέρ αυτής της υποψηφίας. Συγγνώμη, το πράσινο κουμπί είναι, ε, κουμπί είναι υπέρ, ε, το κόκκινο κατά, υπέρ το πράσινο κατά το κόκκινο κουμπί και οι εποχές λευκό. sorry. This is the test. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δοκιμαστική, όπως σας είπα, μυστική ψηφοφορία. Οπότε απλώς δοκιμάζουμε το μηχάνημα. Έχουμε υπεράριθμο στο ΕΛΚ. Δύο. Ένας. Εντάξει τώρα. Οπότε αφήστε τις κάρτες μέσα στο μηχάνημα. Εντάξει, εξοικειωθήκατε με τα μηχανήματα. Τώρα περνάμε στην κανονική ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο μηχάνημα που δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέπω ότι έχει νερό στο μηχάνημα και δεν ε, μπορώ να βάλω την κάρτα μου. Υπάρχει κάποιος τεχνικός ή μπορείτε να αλλάξετε θέση για να δούμε αν εκεί λειτουργεί η κάρτα σας. Yeah, it's working. Okay, then can I... Εντάξει τώρα, οπότε κηρύσω την έναρξη της ηλεκτρονικής μυστικής ψηφοφορίας για τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Have you all Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Οπότε εξελέγει με 38 ψήφους η κυρία Νικόλ Σόνοβα. Συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε. Ελάτε εδώ στο Προεδρείο να λάβετε τη θέση σας. Ελάτε να κάνουμε χειραψία και θα προεδρεύσετε εσείς τις ψηφοφορίες για τους τέσσερις αντιπρόεδρους. So, thank you. Ευχαριστώ πολύ που με εμπιστευθήκατε. Τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να πω λίγα λόγια γιατί εξελέγην, αλλά δεν τα έχω ετοιμάσει γιατί σήμερα το πρωί το έμαθα. Όχι και ιδιαίτερα νωρίς. Τώρα πρέπει να ακυρώσω τις διακοπές που είχα προγραμματίσει με τον σύζυγό μου και αυτό θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου το κάνατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Είμαι από τη Σλοβακία. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν ε, να μιλήσω σλοβακικά για να ακούσετε την ωραία γλώσσα. Αλλά μετά θα μιλάω αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου η οποία με πρότεινε για αυτή τη θέση. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ξέρω πως δεν ήταν εύκολη η κατάσταση. Καταρχάς, να σας περιγράψω ποια είμαι. Ποιαν εκλέξατε ως πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης. Από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική, ασχολούμαι με τα κοινωνικά θέματα. Το 2010-2012 ήμουν ε, υφυπουργό στο Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων, όπου ασχολήθηκα με τα θέματα αυτά, τα οποία μας απασχολούν και εδώ, στην Επιτροπή αυτή. Πρώτα απ' όλα, κυρίως, Ασχολήθηκα με άτομα με πνευματική ή σωματική αναπηρία και με την κοινότητα των Ρωμά. Είναι μια μεγάλη μειονότητα στην Σλοβακία. Μισό εκατομμύριο. Εκ των οποίων οι περισσότεροι ζουν σε συνθήκες που δεν αρμόζουν στον 21ο αιώνα. Επεξεργάστηκα μια στρατηγική για την ένταξη των ατόμων αυτών στην σλοβακική κοινωνία. Πέρα από την εκπαίδευση ασχολήθηκα κυρίως με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Να μην εξαρτώνται από κρατικά επιδόματα. Ασχολήθηκα λοιπόν όπως είπα πολύ και με τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Θέλω και η Επιτροπή μας να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Είμαι ένα άτομο που με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη πρακτική δράση δεν θέλω απλώς ε, να κάνω πολιτικές διακηρύξεις. Με ενδιαφέρει η πράξη. Θεωρώ ότι η Επιτροπή αυτή είναι η σημαντικότερη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα ήθελα όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τις μικροκομματικές ε, αντιπαραθέσεις όπως τις βλέπουμε στην Ολομέλεια. Ε, εκεί μπορεί να έχουν τη θέση τους, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει να ασχολούμεθα με πολύ συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή με βάση στοιχεία να συζητούμε και να αποφασίζουμε μόνο με συγκεκριμένα στοιχεία μπορούμε να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα οι πολιτικές διακηρύξεις δεν βοηθάνε. Η Επιτροπή αυτή ασχολείται απευθείας και θέλει να επηρεάσει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Είμαι άτομο που ενδιαφέρομαι για την επίτευξη συνένεσης και συμβιβασμών. Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή για να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη σας. Δεν ήταν εύκολο να ε, εκλέξετε κάποιον για τον οποίο δεν ξέρετε τίποτα. Και επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου προς την ομάδα μου, την ομάδα ECR των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και ιδιαίτερα την κυρία Σύντο και την κυρία Ραφάλσκη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ μόνιμος πρόεδρος ε, να αναλάβω τις ευθύνες, χρειαζόμαστε και τους αντιπρόεδρους. Οπότε σας παρακαλώ ε, προτάσεις για αντιπροέδρους. Κυρία Γιονγκέρους, για πρώτο αντιπρόεδρο από πλευράς των σοσιαλιστών, την κυρία Βίλνια Μπλίνκοβιτσίε. Λοιπόν, αποδέχεστε την υποψηφιότητα. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Λοιπόν, για τη θέση δεύτερο αντιπρόεδρο. Δεν βλέπω την κάρτα σας, αλλά πείτε μου. Βίλιαμσον. Ευχαριστώ πολύ. Για δεύτερο αντιπρόεδρο η φίλη μου εδώ δεξιά μου, η κυρία Σάντρα Περέιρα. Έχει μεγάλη εμπειρία, δουλειά στα συνδικάτα και έχει αφιερωθεί στα κοινωνικά θέματα. Θα είναι θαυμάσια αντιπρόεδρος για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Κυρία Σάντρα Περέιρα, την αποδέχεστε την υποψηφιότητα. Ναι, την αποδέχομαι. Ωραία. Οπότε τι λέτε κι εσείς. So we have the... Ωραία, έχουμε και δεύτερη αντιπρόεδρο. Τώρα για την θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Παρακαλώ, κύριε Κάζα. Ναι. Τον κύριο Τόμας Ζεντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Στεχόφσκι. Δέχεστε. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Και για την θέση τετάρτου αντιπρόεδρου. Η πράσινη, παρακαλώ. Ναι. Στην κυρία Λάγκεντζίντερ, θέλω να προτείνω. Λάγκεντζίμπεν, κυρία Λάγκεντζίμπεν, δέχεστε, δέχεστε. Ωραία. Congratulations. Συγχαίρω και, και Έχουμε λοιπόν τους τέσσερις αντιπρόεδρους και μπορούμε να αρχίσουμε την εργασία μας. Okay, so it's the end of the... Ωραία. Λοιπόν, κλείνω τη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Okay.